στην ιστοσελίδα ε, η Ολομέλεια Απευθεία θα δείτε ε, το σχετικό τίτλο που έχουμε δημοσιεύσει για τα πρακτικά αυτή τη συνεδρίαση. Στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού μας υπογράψαμε τέσσερις πράξεις σχετικά με την νομοθετική διαδικασία και οι τίτλοι αυτών των πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδριάς.